Λοιπόν, ξεκινάμε τις εργασίες μας και <clears throat> ξεκινάμε με την έκθεση της κυρίας Τζαβέλα. Παρακαλώ λοιπόν να καθίσετε διότι έχουμε καθυστερήσει. Λοιπόν, καθίστε σας παρακαλώ. Και ησυχία για να δώσουμε το λόγο στην συνάδελφο κυρία Τζαβέλα και έχουμε 30 λεπτά για αυτή τη συζήτηση. Παρακαλώ λοιπόν, σας παρακαλώ. Αρχικά θα ήθελα να χαιρετήσω τη νέα στρατηγική της Επιτροπής για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική αυτή εντάσσει την ανάπτυξη των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 στο πλαίσιο της έξυπνης, βιώσιμης και περιεκτικής ανάπτυξης. Η γνωμοδότηση. Πρώτον, ζητά την καλύτερη ενσωμάτωση των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών στην Ένωση. Ζητά την προσαρμογή της πολιτικής συνοχής στα δεδομένα των απομακρυσμένων περιφερειών στους τομείς που αφορούν την Επιτροπή μας, δηλαδή στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, των ΜΜΕ και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Δεύτερον, η γνωμοδότηση επισημαίνει ότι οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο γέφυρας γνώσης μεταξύ Ευρώπης και τρίτων χωρών και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να συνυπολογίζουν το σημαντικό ρόλο των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών στο πλαίσιο των επαφών με τρίτες χώρες. Τρίτον, κλιματική αλλαγή. Πρέπει να συμπεριληφθούν ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές στο πλαίσιο στρατηγικής της Ένωσης για τις κλιματικές αλλαγές, δεδομένου ότι είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στην άνοδο της στάθμης των υδάτων. Και τέταρτο, η γνωμοδότηση ε, αναφορικά, η ε, αναφορικά με το διαδίκτυο και την πρόσβαση επισημαίνει ότι η ψηφιακή οικονομία προωθείται ως ένα από τα εργαλεία που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να βγει από την κρίση. Επομένως, οφείλουμε να αποδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωση των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Συμφωνούμε με τις προτάσεις που υπάρχουν στην έκθεση για το ψηφιακό θεματολόγιο Del Castillo Report που καταγράφεται ότι οι ασύρματες τεχνολογίες περιλαμβανομένης και της δορυφορικής θα μπορούσαν να παράσχουν στους πολίτες των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών, άμεση και παντού πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο. Τέλος, κύριε Πρόεδρος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, των οποίων οι χώρες ε, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις απομακρυσμένες αυτές περιοχές. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν αυτούς τους συναδέλφους και όλους οι οποίοι συνέβαλαν στην γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Τζαβέλα και τώρα το λόγο έχει, έχουν ισχυώδει οι και ξεκινώ με τον κύριο Βανίστελ Ρόι. Εσείς έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ εξισορροπημένη η έκθεση μας έχετε παρουσιάσει πολύ καλά την άποψή σας, όμως θα ήθελα μερικά ζητήματα να θέσω. Πρώτον, Δεν χρειάζεται να αμφιβάλλουμε για τη θέση των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ενισχύθηκε η θέση τους ε, στη συνθήκη της Λισαβόνας, αν δει κανείς ε, άλλες περιφέρειες και την επιπλέον χρηματοδότηση παραμένουν στο ίδιο επίπεδο, άρα δεν βλέπω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει ε, διατηρηθεί η θέση τους και επίσης ε, γνωρίζετε ότι οι ιδιαίτερα απομακρυσμένε περιφέρειες έχουν πολύ καλή επικοινωνία και επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό, αλλά έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η στρατηγική 2020 δίνει νέες δυνατότητες, δίνει νέες ευκαιρίες Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει κανείς μόνο τα ευρύτερα ζητήματα που επηρεάζουν ιδιαίτερα τα νησιά, αλλά πρέπει να εξειδικευτούμε σε μερικές ε, περιφέρειες και θα ήθελα να δούμε λίγο περισσότερα πράγματα. Υπάρχει μια ευφυής ε, εξειδίκευση. Μπορεί να πάει κανείς στα νησιά και να τους ρωτήσει τι ακριβώς κάνετε ιδιαίτερα καλά, γιατί τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπόδειγμα. Η Γαλλική Γουιάννα, για παράδειγμα. Εκεί αρχίσαμε τους δορυφόρους του Γαλιλαίου, για παράδειγμα. Ε, όλη, ε, όλη η προσοχή έχει στραφεί εκεί και αυτό τους δίνει ε, τους δίνει, τους δίνει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες. Ε, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε με τις υπόλοιπες ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, γιατί βρίσκονται γεωγραφικώς σε μια καλή θέση για να μας δώσουν για να αξιοποιήσουν ιδιαίτερες ευκαιρίες όσον αφορά λοιπόν την υποδομή, τις επενδύσεις ε, και, τους, ε, και την έρευνα μπορούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτές τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, ε, να βελτιώσουμε την εικόνα τους, να προσελκύσουμε σε αυτές μεγαλύτερη προσοχή και να μεταφέρουμε και ερευνητικέ δραστηριότητε εκεί, για παράδειγμα, όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή. Αυτό θα ήθελα μόνο να προσθεθεί στο κείμενο. μπορούμε να ρωτήσουμε τις περιοχές αυτές σε τι εξειδικεύονται, ώστε όταν ε, κάνουμε μεγάλες ε, επενδύσεις για υποδομές στις ε, περιοχές αυτές, να μπορούν να υποφεληθούν σωστά. Και όσον αφορά τα flagships, νομίζω ότι τα προγράμματα αυτά όταν βλέπουμε για παράδειγμα την έρευνα, την ανάπτυξη, τα προγράμματα που πρέπει να εφαρμοστούν στο μέλλον και πάλι μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο οι περιφέρειες αυτές. Πρέπει να συμμετέχουν στα προγράμματα flagships, να ζητήσουμε να υπάρχει συγκεκριμένη παράγραφος στα προγράμματα αυτά που θα ε, αφιερώνεται στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες. Αυτά είναι τα σχόλια που θα ήθελα να κάνω και θα αναφέρονται και στις ε, τροπολογίες που θα υποβάλω. Ευχαριστώ πολύ. Ehm. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι σκιώδης ε, για αυτήν την έκθεση για αυτό το θέμα αλλά θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στις άλλες σκιώδης η κυρία Τάκουλα κάποιος την αντικαθιστά όχι ο κύριος Τούρμες ε, ε, επίσης απουσιάζει κάποιος άλλος θέλει να πέμβει υπέρ των πρασίνων ο κύριος Τσέτσεστερ τότε μπορώ εγώ να μιλήσω ίσως σαν σκιώδης για αυτό το θέμα και συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Βανίστελ Ρόι διότι πιστεύω ότι η σημασία που πρέπει να δοθεί σε αυτές τις άκρα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η προοπτική αυτή λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθεί με τις πολιτικές οι οποίες ε, είναι αφιερωμένες η έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών αναφέρεται και στις πολιτικές ε, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε φορολογικά, τελωνιακά ζητήματα, αλλά φυσικά και πολλά θέματα τα οποία απέφεραν καρπούς, αλλά αυτό που είναι εξίσου σημαντικά σήμερα ε, σε σχέση με το στόχο της υπερίληψης αυτών των εξόχως απομακρυσμένων περιοχών οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμπερίληψή τους στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να δράσουμε ε, στην επίθεση, να προτείνουμε, να δώσουμε προκλήσεις ώστε να δώσουμε αξία σε αυτές τις ιδιαιτερότητες που έχουν αυτές οι περιοχές, γεωγραφικές, δαφικές αλλά και μορφολογίες που είναι σημαντικές για να δούμε ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που μπορούν να βοηθήσουν για την Ευρώπη του 2020. Για παράδειγμα, το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Είναι ένα σημαντικό χαρτί που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιοχέ που έχουν συγκεκριμένα μορφολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά και από την αδυναμία της ε, ενεργειακής εξάρτησης να γίνουν ένα ισχυρό σημείο για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Και θεωρώ ότι ε, πέραν από τα ad hoc προγράμματα θα πρέπει να δράσουμε ως προς την προσαρμογή στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων των βασικών προγραμμάτων για να επιτύχουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020. Αναφέρθηκα στο θέμα της ενέργειας αλλά υπάρχει και το θέμα του κλίματος το οποίο είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη και η συγγήτρια η κυρία Τζαβέλα το υπενθυμίζει. Είναι επίσης σημαντικό και το θέμα της έρευνας. Πώς μπορούμε εμείς, με ποια μέσα να ε, βοηθήσουμε ε, σε ιδιωτερότητες που έχουν αυτές οι περιοχές, να ξεπεράσουμε τις αδονομίες και να δώσουμε αξία στις ιδιωτερότητες τους. Ακόμα και στον τομέα της έρευνας λοιπόν, να δούμε πού βρίσκονται τα ισχυρά σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και να προσαρμόσουμε το γενικό πρόγραμμα σε αυτό το στόχο της συμπερίληψη, της ενσωμάτωσης αυτών των εξόχων απομακρυσμένων περιφερειών ε, με περισσότερο ομοιόμορφο τρόπο και με λιγότερες διαφορές και καθυστερήσει. Το πρόγραμμα τη έρευνα είναι ζωτική σημασία και εμείς οι οποίοι είμαστε αυτοί που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, ε, η κυρία Μαντουρέλ είναι συγγήτρια για το θέμα αυτό, αλλά και όλοι θα πρέπει να ενσωματώσουμε και αυτό το στόχο στα βασικά γενικά προγράμματα της έρευνας. Ένα άλλο θυμίο το οποίο υπενθυμίζει η συντάκτρια κυρία Τζαβέλα είναι το θέμα των επικοινωνιών, το να μπορέσουμε να επιτύχουμε στόχους ε, ψηφιακούς ε, και ψηφιακής ενσωμάτωσης σε αυτές τις περιοχές είναι η δυνατότητα να του προσφέρουμε μεγάλη στήριξη και για την οικονομία τους και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στις περιοχές αυτές. Επομένως, η προσέγγιση η οποία υπενθυμίστηκε, ε, η πρόταση που γίνεται να προσέξουμε αυτές τις περιοχές, που σημαίνει ότι να ε, χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες της εναλλακτικές λύσεις της εξειδίκευσης, ίσως είναι η καλύτερη λύση για να επιτύχουμε το στόχο της ενσωμάτωσης, της ένταξης και μιας ε, πιο συνεκτικής πολιτικής. Και η ομάδα μου λοιπόν θα καταθέσει τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση, συνεργαζόμενοι και με τους συναδέλφους που προέρχονται από αυτές τις περιοχές και γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμά τις ιδιαιτερότητές τους και να συνεργαστούν μαζί μας λοιπόν για να επιτύχουμε αυτό το στόχο της ένταξης. Δεν είναι εδώ παρόντες οι άλλοι τι συζητητές και θα δώσω λοιπόν το λόγο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω να κάνω μία παρέμβαση διότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζητήσουμε μία καλύτερη ένταξη όλων των περιοχών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασχέτως ε, των, ε, της γραφικής του θέσεως αλλά γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία με τις χώρες διότι υπάρχουν δυσλειτουργίες υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι απομακρυσμένες και φτωχές και πληρώνουν τα τρόφιμα πολύ πιο ακριβά από ότι το κέντρο και αυτοί οι οποίοι εμπορεύονται τα τρόφιμα έχουν διαφορετική άποψη και θα μπορούσε η Ευρώπη με τη βοήθειά της να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσει του πληθυσμού και να δημιουργήσει μία γέφυρα κατά τρόπον ώστε να υπάρχουν συνεργασίες για να ανταποκριθεί καλύτερα κανείς στις ανάγκες των χωρών και να τους επιτρέψει να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωή τους. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ εις ε, τις επιπτώσεις των κλιματολογικών ε, λαγών, την άνοδο των υδάτων για να μπορέσουμε ε, να προβλέψουμε τις μελλοντικές εξελίξεις όσο δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Επομένως, να δώσω το λόγο στην Άννα Λουτσία Πίντο, η οποία είναι συντονίστρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα που σχετίζονται με τις περιοχές αυτές. Παρακαλώ, κυρία Πίντο. Καλημέρα σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χαιρετίζει την γνωμοδότηση της ΙΤΡΕ ε, και θεωρεί ότι αυτές, ε, αυτά τα μέτρα προσπαθούν να απαντήσουν στις ανάγκες σύμφωνα με τα <coughs> με το σχετικά άρθρα των συνθήκων και ε, υπάρχουν ιδιαίτερες διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν μία ανάκαμψη των περιοχών αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τις επιπτώσεις της κλιματολογικής αλλαγής επί της ανταγωνιστικότητας των χωρών και ε, πρέπει να περιληφθούν ε, τα μέτρα για την ε, έρευνα στις ε, προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2018 κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί η οικονομία και να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε ελάχιστο χρόνο, αλλά η κυρία Τζαβέλα θα μπορούσε να απαντήσει εντός λίγων λεπτών, παρακαλώ κυρία Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ όλους για τις προτάσεις τις οποίες κάνατε. Θα περιμένω τις ε, τροπολογίες τις οποίες θα καταθέσετε και ελπίζω ότι θα βγούμε με μία γνωμοδότηση η οποία θα είναι προς όφελος των ε, πολιτών των απομακρυσμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από τη συζήτηση λοιπόν, κατάθεση τροπολογιών μέχρι την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ο λόγος στην κυρία Κρόιτσμαν, η οποία αντικαθιστά τον ε, Μάικολ Τέρερ. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να παρουσιαστώ. Είμαι από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και τώρα βρίσκομαι εδώ σε μια σημαντική επιτροπή καθότι ανταλλάξαμε θέσεις και ο κύριος Τόιρερ με παρεκάλεσε να αναλάβω την έκθεσή του στην Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ενεργείας πράγμα το οποίο έπραξα με μεγάλη ευχαρίστηση γιατί πιστεύω ότι ότι η ελκυστικότητα της Ευρώπης είναι πολύ βασικό θέμα. Πρέπει να ενισχύσουμε τη βιομηχανία μας και γι' αυτό θα συμφωνήσετε φαντάζομαι με τις προτάσεις που διατύπωσα. Βεβαίως υπάρχουν ακόμη, υπάρχει ακόμη χρόνος να υποβάλει κανείς τροπολογίες. Έχουμε ε, καταρχήν διάφορα βασικά θέματα την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς διότι πρέπει να προσελκύσουμε επενδύσεις στην Ευρώπη και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μία κατάργηση της γραφειοκρατίας και περιορισμό των διατάξεων διότι η Ευρώπη έχει τον, τη μεγαλύτερη εσωτερική αγορά στον κόσμο πράγμα το οποίο είναι μεγάλο προσόν για τις επιχειρήσεις και πρέπει να την ενισχύσουμε για να αναπτυχθεί περαιτέρω. Πουθενά αλλού δεν μπορεί κανείς ε, να διαθέσει τις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σε μία τόσο μεγάλη αγορά και ε, πρέπει να μπορεί κανείς να υποφεληθεί από μία βελτίωση της ανταγωνιστικότητος και της αποτελεσματικότητος. Για να υπάρχει όμως αυτό χρειαζόμαστε μία ενιαία αντιμετώπιση και ρυθμίσεις διότι διαφορετικά τα προγράμματα δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Φροντίζουμε λοιπόν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να δημιουργούν θέσεις εργασίας στο μέλλον οι οποίες θα οδηγούν σε εξειδίκευση των ρόλων και σε αριστεία. Στο χώρο δε αυτό υπάρχουν ακόμη μεγάλες δυνατότητες βελτιώτης. Ε, παραδείγματος χάρη αν συγκρίνουμε την ισχύουσα, το ισχύον επίπεδο της ε, βλέπουμε ότι στην Ευρώπη ε, ε, εάν εξετάσουμε το μέσο όρο και το συγκρίνουμε ε, με τη Γερμανία βλέπουμε ότι οι πολλές έρευνες μετακινούνται από την Ευρώπη στην Αμερική όπου παραδείγματος χάρη διατηρούν την έρευνα στον τομέα της γενετικής τεχνολογίας ενώ στην Ευρώπη δεν προωθείται. Ε, υπάρχουν βέβαια διάφορες δυνατότητες ε, για συνεργασίες και δεν πρέπει ε, να υποτιμά κανείς τις δυνατότητες αυτών των συνεργασιών και να το συζητήσουμε διότι πέραν αυτού πρέπει να προωθήσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του πρόοδου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι υποτιμούμε την ε, ε, καινοτόμα δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διότι τα ποσοστά ε, που, της αγοράς που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προχωρήσουν πιο αποτελεσματικά για να υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση win-win θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη βάση έρευνας και να μην εστιαζόμαστε μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στον ερευνητικό τομέα για να μπορέσει η Ευρώπη να διατηρήσει και να επενδύσει σε ε, υποδομές διεθνούς επίπεδου όπως η τεχνολογία και ε, η βιομηχανία και θα πρέπει να επιλύσουμε και το θέμα της μεταφοράς της ενεργείας διότι η ενέργεια είναι ένας τομέας κλειδί για να ε, δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στην Ευρώπη αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε ε, την τιμή της ενεργείας για να μην διακινδυνεύει ο τομέας της βιομηχανίας υπάρχουν συνεχείς αυξήσεις ε, της τιμής ενεργείας και αυτό υποβιβάζει το βιομηχανικό επίπεδο της Ευρώπης. Θα πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε χωρίς περαιτέρω αυξήσεις των τιμών ενεργείας. Χρειαζόμαστε έξυπνες λύσεις γιατί ο καθένας θέλει να περιορίσει το διοξίδιο του άνθρακος το οποίο είναι διαμφισβήτητο αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια ισορροπία χωρίς να αυξάνουμε τόσο πολύ τις τιμές ενεργείας ώστε να είναι εις βάρος των επιχειρήσεων της Ευρώπης και ιδίως των μικρομεσαίων οι οποίες ε, πλήττονται περισσότερα. Θα προσπαθήσω δηλαδή να ε, προσθέσω και νέες ιδέες στην έκθεση του συναδέλφου Τόιρετ και περιμένουμε τα μεγάλο ενδιαφέροντος τα σχόλια των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ κύριε Κρόιτσμαν. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε 17 λεπτά στη διάθεσή μας γιατί μετά έρχεται ο Υπουργός Έστεγκαρτ και επομένως δεν έχουμε πολύ χρόνο για να το συζητήσουμε. Να δώσω το λόγο στον κύριο Κέλλη, ο οποίος είναι σκιώδη συντάκτης για το εκ μέρους του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και τον κύριο Κρόιτσμαν ε, για τα εισαγωγικά του σχόλια. Είναι προφανώς ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρώπη, ειδικότερα εν μέσω μιας κρίσης. Πρέπει να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση, πρέπει να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Και βέβαια το να, επενδύσουμε, να υπάρχουν επενδύσεις στην Ευρώπη είναι ουσιαστική σημασία. Υπάρχουν κάποιοι τομεί ε, στην ε, Ευρώπη Εντάξει, όχι πάρα πολλοί, αλλά είναι αρκετοί, για τους οποίους ε, χάνουμε έδαφος σε σχέση με την Κίνα και πρέπει να έχουμε μια συνολική στρατηγική ε, ανάπτυξης ε, ε, στην Ευρώπη, ώστε τουλάχιστον να φτάσουμε στο 26% του FDI Έχουμε επαναχωρήσει τα τελευταία χρόνια. Ελπίζω να φτάσουμε και πάλι στο 26% και αν το κάνουμε αυτό θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πολλές θέσεις απασχόλησης. Τα σημεία ε, που είναι επίσης πολύ σημαντικά είναι οι συνδέσεις μεταφορών, όπως για παράδειγμα οι σιδηροδρομικές συνδέσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα των φορολογικών συνθήκων, ε, ε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ε, τα θέματα του ορίζοντα 2020 πρέπει να είναι κατάλληλα σε σχέση με τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε, να είναι ευθυγραμμισμένα με την αγορά. Η έρευνα πρέπει να ακολουθεί να οδηγεί σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης Για παράδειγμα, ε, η παραγωγή ε, οθονών ε, τηλεοπτικών ε, flat screen ε, δεν γίνεται πια σχεδόν καθόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα δείγμα. Το θέμα της ευρυζωνικής, του ευρυζωνικού διαδικτύου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικότερα σε σχέση με τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, πράγμα το οποίο επίσης συζητήσαμε προηγουμένως. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις και πρέπει να δείξουμε ότι θέλουμε να τις βοηθήσουμε όπως και άλλους τομείς να συμμετέχουν σε αυτή την ανάπτυξη της ε, Ευρώπης. Υπάρχει και το θέμα της επιμελητίας. Είναι σημαντικό για όσους επενδύουν στην Ευρώπη η σταθερότητα του πολιτικού και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, όπως επίσης και η δομή των τηλεπικοινωνιών. Αυτά είναι βασικοί τομείς. Αν μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας σε αυτούς τους τομείς, τότε ε, θα βελτιωθούν και οι επενδύσεις και μπορούμε πραγματικά να αναπτυχθούμε πολύ ως προς αυτούς τους τομείς. Ε, Παρίσι, Λονδίνο, Φραγκφούρτη τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά ε, και άλλες πόλεις ε, έχουν βελτιωθεί πολύ. Πρέπει να μάθουμε από τις πόλεις αυτές και να ε, εξασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις είναι στο σύνολο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους του 2020. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Ο κύριος Κορέιρα Κάμπος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας συγχαρώ και για την εκλογή σας, αλλά θα ήθελα να συγχαρώ και τον συνάδελφο Κρόιτσμαν, που είναι πλέον στην Επιτροπή μας. Τον γνωρίζουμε από την δουλειά του στην Επιτροπή Εστερικής Αγοράς. Ευχαριστούμε και τον κύριο Τερέρ βέβαια αλλά θα ήθελα να κάνω και μερικά σχόλια. Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με αυτές τις πέντε παραγράφους, αλλά έχουμε και κάποιες προτάσεις που θα θέλαμε να προσθεθούν. Η πρώτη πρόταση, το ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτήν ε, την ε, θετική ανταγωνιστική πτυχή του ανθρώπινου δυναμικού μας, ε, να μην ε, το αφήσουμε σε χειμερή ανάρκη. Έχουμε επίσης και το θέμα της κατάρτισης, ε, της εκπαίδευσης ε, στην Ευρώπη που συνδέεται με την καινοτομία. Τα πανεπιστήμια πρέπει να συνδέονται περισσότερο με τα τεχνολογικά ιδρύματα και γενικότερα με την έρευνα. Είναι μια σιωπηρή δουλειά η οποία όμως πρέπει κάπως να αξιολογηθεί. Η τυποποίηση επίσης ε, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό θέμα επί του οποίου θέλουμε να ε, αναπτύξουμε τις βιομηχανικές πτυχές στην Ευρώπη ε, είναι σημαντική η στόχη στο πλαίσιο του 2020 όσον αφορά την αηφορία, την ενεργειακή, την κλιματική μεταβολή και όλα αυτά τα πράγματα που συζητήσαμε και χθε, ε, την ενέργεια του ε, ανεφοδιασμού ε, σε τρόφιμα αλλά και σε νερό, η ιατρική, η, όλα τα, όλες οι βιολογικές πτυχές, η πράσινη τεχνολογία και ο κατάλογος δεν σταματάει εδώ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε και τη βασική μας βιομηχανία όπως... Ε, τα διαστημικά, ε, την ε, φαρμακοβιομηχανία. Δεν είναι δυνατόν να τα ξεχάσουμε αυτά και να τα αφήσουμε απλώς να πεθάνουν. Λίγο όμως τους αναφέρουμε αυτούς τους βασικούς τομείς της βιομηχανίας μας. Είναι σημαντικό τμήμα όμως της ανταγωνιστικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να τις ε, αναφέρουμε, όπως πολύ σημαντικός είναι και ο τουρισμός. Δεν πρέπει να υπάρχουν πλέον εμπόδια στην εσωτερική αγορά, εξακολουθούν να υφίστανται. Υπάρχει το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου που πρέπει να ενισχυθεί. Οι χρηματοοικονομικές ε, υπηρεσίες ε, πρέπει να επενδύσουμε σε μια διατλαντική συνεργασία, γιατί είναι πραγματικά μια πηγή έμπνευση για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, για παράδειγμα, τις πτωχεύσεις ένα μόνο, μια μόνο επίκριση στο σημείο 3 όταν μιλάμε για τη μείωση των, ε, ε, του κόστους για τις επιχειρήσεις, το business cost, ε, εγώ θα προτιμούσα να έχουμε μια θετική διατύπωση, δηλαδή να μιλήσουμε για αύξηση του ωφέλους. Και τέλος, όπως είπε και άλλος συνάδελφος, ε, πρέπει να δούμε και την εξέλιξη του ε, κρατικού χρέους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά έχουν ε, αντίκτυπο στις επενδύσεις. Εντάξει, είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ θετικά τα πράγματα αλλά δεν είναι δυνατόν να το αγνοούμε απλώ επειδή είναι αρνητικό, ειδικά σε μια τέτοια γνωμοδότηση. Ευχαριστώ τον κύριο Κορέιντα Δεκάμπο. Τώρα, σε πέντε λεπτά στι 11.30 θα έρθει ο Υπουργό. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μου. Έχω τρει παρεμβάσει μετά από την, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά το συντάκτη τη γνωμοδότηση. Θα προσπαθήσω να σα καλύψω όλου. Ο κύριο Πρόντι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. φρονώ ότι πριν εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό θα πρέπει να ε, κυριαρχήσει το εξής. Η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει κατασκευαστική δραστηριότητα. Και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσουμε και από εκεί και πέρα έρχονται συνέπειες. Έχουμε ένα βιομηχανικό κατασκευαστικό τομέα ο οποίος ε, κυριάρχησε, είχε προεξάρχοντα ρόλο σε όλο τον πλανήτη και δεν μπορούμε αυτή ε, την βιομηχανική πολιτική να την εγκαταλείψουμε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική που θα διευκολύνει τις επενδύσεις και στην Ευρώπη και θα ασχοληθεί και με το θέμα της ανταγωνιστικότητας, η οποία θα πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ενώπιον των υπολείπων. Να σας δώσω το παράδειγμα της Κίνας. Η Κίνα έχει κάποιες πτυχές της πολιτικής της, στην οποία προφανώς θέλει να γίνει ε, ο κατασκευαστής του κόσμου. Αυτό δεν είναι δυνατόν, διότι δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε εμείς και δεν μπορεί να το εγγυηθεί και η Κίνα. Δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υπάρχει συνεχής ε, κατασκευή όπως ακριβώς θέλει να ε, θεωρεί η ίδια ότι έχει και γιατί υπάρχουν ε, οικονομικές κρίσεις αλλά και δημογραφικές κρίσεις στην Κίνα. Επομένως, θα πρέπει να ορίσουμε το πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τουλάχιστον τον παραγωγικό ιστό, ο οποίος είναι ζωτική σημασία για την επιβίωσή της. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι σε κάποια χρόνια, σε μια δεκαετία, όπως ακριβώς συνέβη και με την Ιαπωνία και με την Κίνα, θα βρεθούμε σε ένα ισότιμο σημείο ανταγωνιστικότητας και θα πρέπει και αυτό να το συμπεριλάβουμε στο λογαριασμό μας. Ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο, ο κύριος Βέμπερ. Ε, είναι κύριος ο Βέμπερ γιατί υπάρχει και μία κυρία Βέμπερ σε δύο λεπτά. Πρέπει να σας πω ότι είμαι αντιπρόεδρος της ε, ε, ε, Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ενώσεως Κίνα όπου υπήρξε μεγάλη εξέλιξη των επενδύσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία πέντε χρόνια και αυτό είναι μόνο η αρχή. Είναι εξαιρετικό από πολλές απόψεις αρχή αυτή η, αυτός ο προγραμματισμός των επενδύσεων από την Κίνα μπορούν, ε, να μπορέσουν να συντονιστούν στην Ευρώπη. Δηλαδή χρειαζόμαστε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διότι η ε, Κίνα παίζουν ε, το κάθε ένα από τα 27 κράτη-μέρη έναντι του άλλου για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Τα, έχουμε πάμε λοιπόν σε άλλους σχηματισμούς αυτές ε, τις ε, μεθόδους. Δηλαδή στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχει μια επιτροπή συντονισμού των ε, αλλοδαπών επενδύσεων η οποία κάθε φορά που παρουσιάζεται μια περίπτωση αξιολογεί την επένδυση αυτή και αξιολογεί πόσο θα βοηθήσει τις αναδυόμενες ε, ή ε, εξελισσόμενες ε, τέτοιες τεχνολογίες. Ο κύριος Ταγιάννη επιθυμεί να υπάρξει κάτι παρεμφερές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι βάσει της αμοιβαιότητος η Κινέζοι ε, έχουν μια πολύ ε, ε, συγκεντρωμένη πολιτική σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν τρεις τομείς. Πάρα πολλούς απαγορευόμενους τομείς που αναφέρεται στις δημόσιες επιχειρήσεις, στις τράπεζες, στις θαλάσσιες μεταφορές και ένα πολύ μακρύ κατάλογο. Ο τομείς όπου υπάρχει ένα, κάποια τροχοπέδη όπως τα αυτοκίνητα, η αυτοκινητοβιομηχανία όπου οι ε, Ευρωπαίοι δεν μπορούν να έχουν πάνω από 49% της επενδύσεως στην Κίνα ενώ οι Κινέζοι μπορούν να αγοράσουν ολόκληρη τη Βόλβο και άλλοι μίσο που οι Κινέζοι χρειάζονται τη τεχνολογία μας πρέπει λοιπόν να μην είμαστε αφελείς στην ε, Επιτροπή, στο στην πολιτική επενδύσεων και να δημιουργήσουμε μια νέα επιτροπή για τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Βαλνίστεροι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι στις επενδύσεις, εφόσον μιλάμε για επενδύσεις, μιλάμε για επενδύσεις στην Ευρώπη και πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος επενδύει περισσότερο στην Ευρώπη, οι Κινέζοι. Αν δούμε λοιπόν ε, τι, ε, ποιοι είναι οι πόροι που ρέουν προς την Ευρώπη αν δω το λιμάνι ε, του Ρότερνταμ το μισό είναι στα χέρια των Κινέζων και ακόμη και αν δεν αναφέρουμε αυτές τις εξελίξεις σημαίνει ότι δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε την έκθεση αυτή στα πλαίσια της διεθνούς εξελίξεως και όπως ελέγχθη υπήρξε μία έκκληση και γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ. Θα υποβάλω μία τροπολογία η οποία θα αποβλέπει στην κατάρτιση μιας πιο επιθετικής αντιμετώπισης γιατί ε, εδώ διακυδεύεται το μέλλον μας. Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε συνεχίσουμε και να αναπτύξουμε την Ευρώπη πρέπει να σκεφτούμε ε, τις ε, κρατικές επιδοτήσεις σε στρατηγικά σημαντικούς τομείς, δηλαδή αν θέλουμε να έχουμε στην Ευρώπη πράγματα που θα είναι αποτελεσματικά μετά από 20 χρόνια θα πρέπει να μην ε, τα αφήσουμε όλα στα χέρια των Κινέζων. Θα πρέπει επιπλέον στον τομέα της έρευνας και των υποδομών να δούμε τι γίνεται διότι αν έχουμε σωστές ε, ε, υποδομές τότε θα προσελκύσουμε επενδυτές ενώ διαφορετικά θα συμβεί το αντίστροφο και μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα ε, σημειώσουν ζημιές πράγμα το οποίο πηγαίνει προς την κακή κατεύθυνση. Παρακαλώ να είσαι εσείς όμως κύριε Σιγητά γιατί ήρθαν οι υπουργοί. Ευχαριστώ θα είμαι σύντομος, ευχαριστώ για τις προτάσεις. Θα πω στην κυρία Ντεκάμπος ότι είναι σωστά, ε, πρέπει να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, θα υπάρξουν τρεις τροποδο... Ε, τροπο επ' αυτού για, θα πρέπει να κοιτάξουμε την παραγωγικότητα όχι μόνο από την πλευρά τη θετική αλλά και από την πλευρά του κόστους και της αποδοτικότητας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα... Α, συγγνώμη, μία τελευταία πληροφορία. Κατάθεση τροπολογιών μέχρι την 3η 31 Ιανουαρίου 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα στη συγκεκριμένη συζήτηση να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο να καλωσερίσουμε τον Υπουργό Οέστεγκαρντ, Υπουργό Έρευνας Καιροτομίας και Ανωτέρας Εκπαίδευσης ο οποίος ασκεί την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ζητούμε συγγνώμη για την ε, μικρή καθυστέρηση και η συζήτηση αυτή θα διαρκέσει μέχρι τις 12.30. Να δώσουμε το λόγο στον Υπουργό. Ένα τέταρτο έχετε περίπου στη διάθεσή σας για να μπορέσουμε στη συνέχεια να σας θέσουμε ερωτήσεις και να απαντήσει ο Υπουργός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργό. και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντάς σας ε, για τη νέα σας θέση ως Προέδρου της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας. Ε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δυνατότητα που μου δίνει να, παρουσιάσει... να παρουσιάσω τις φιλοδοξίες της Δανικής Προεδρίας για την έρευνα και την καινοτομία. Από την τελευταία Δανική Προεδρία έχουν γίνει πάρα πολλά και στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θυμάμαι τη σύνοδο στην Κοπενχάγη του 2012 που ελήφθη η απόφαση για την ε, ε, προσχώρηση 10 ε, νέων μελών για τη μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα επίσης είναι μια ιστορική περίοδο στην, για την ευρωπαϊκή ιστορία, όμως είναι διαφορετικός ο κοινός παρονομαστής. Σήμερα υπάρχει μια ε, πολύ έντονη οικονομική κρίση που κλονίζει στη θέμελα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ε, εξέλθουμε της κρίσης αυτής, της οικονομικής κρίσης και παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αφιερώσει προσπάθειες για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων για το κλίμα, την ενέργεια, το περιβάλλον και την ασφάλεια. Και βάσει αυτών η Δανική Προεδρία έχει τέσσερα σημεία εστίαση. Πρώτον, χρειαζόμαστε μία ε, υπεύθυνη Ευρώπη. Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την Ευρώπη ε, είναι να υπάρχει μία βιώσιμη οικονομική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Ένωση, γιατί αυτό δημιουργεί εμπιστοσύνη από τι αγορέ και είναι και βάση ευημερία. Έχουμε ένα άνευ παραλλήλου πλαίσιο, την κοινωνική μέθοδο που μα δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τα τα πρότυπα ε, δικαιοσύνης ε, χωρίς να μειώνουμε την διαφορετικότητα των κοινοτήτων και των πολιτισμών. Ένα βασικό στοιχείο κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας είναι η διαπραγμάτευση του πολιετούς ε, ε, ε οικονομικού πλαισίου που θα, μας, ε, θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε εις πέρας όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεύτερη προτεραιότητά μας είναι η δυναμική Ευρώπη. Ε, ακρογωνιαίος λήθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενιαία αγορά που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και ευημερία για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αγορά αυτή πρέπει να ενισχυθεί, πρέπει καινοτόμε λύσεις να προωθούν οι προκλήσει είναι μεγάλες, η ανάπτυξη είναι χαμηλή, το χρέο είναι υψηλό και ε, χάνονται θέσει απασχόληση. Η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόληση χρειάζονται ενίσχυση. Η ενίσχυση τη αηφόρου ανάπτυξης ε, σημαίνει ενίσχυση ε, της άριστης έρευνας ε, και την ενίσχυση της ε, ανώτατης παιδείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενίσχυση του τριγώνου της ε, γνώσης και επενδύσεις όσο το δυνατόν πιο άμεσες. Δεν θα έπρεπε να είναι ένα μουσείο η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να είμαστε δυναμικοί και να έχουμε πέρα από τα σύνορά μας ισχύ. Τρίτη προτεραιότητα της Δανικής Προεδρίας είναι η πράσινη Ευρώπη. Ε, πρέπει να είμαστε στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας ηγέτες. Πρέπει να μπορούμε να προσαρμοστούμε σε μια πιο πράσινη κοινωνία, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις για την έλλειψη πόρων, την μόλυνση και τις κλιματικές αλλαγές. Η έρευνα και η ανάπτυξη στους τομείς αυτούς πρέπει να ενισχυθεί συνεπώς. Και αυτό θα, οδηγηθεί, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και σε νέες θέσεις απασχόλησης, γιατί η κατανάλωση θα αυξηθεί κατά ένα τρίτο κατά τους επόμενους, ε, κατά 25, επόμενα 25 χρόνια και ε, οι πόροι όλο και μειώνονται. Η ενεργειακή αποδοτικότητα μπορεί να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια ευρώ ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να επενδυθούν τα ποσά αυτά στην ανάπτυξη και τι πράσινε θέσει απασχόληση εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε αυτό να δημιουργήσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Ε, χρειαζόμαστε και μια ασφαλή Ευρώπη και ο καλύτερο τρόπο για να το επιτύχουμε αυτό, την ασφάλεια των πολιτών, των είναι ε, σε έναν παγκοσμιούμενο κόσμο πιο συντονισμένες προσπάθειες και ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία. Εκτός λοιπόν από το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, το βασικό πλαίσιο της Προεδρία μας θα είναι η παρακολούθηση των στόχων για το 2020. το ε, πρόγραμμα Horizon 2020 είναι ο βασικός, η βασική πολιτική κινητήρια ε, δύναμη προς την κατεύθυνση αυτή. Το Συμβούλιο κατά την Προεδρία μας θα έχει να αντιμετωπίσει βασικές νομοθετικές ε, προτάσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης ε, και της καινοτομίας, συγγνώμη, τον ορίζοντα 2020, την στρατηγική ατζέντα για την καινοτομία, για το GMES και για την Ευρατόμ το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από την επιστήμη και την καινοτομία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ορθώς ε, ενισχύει το επόμενο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας και τον ορίζοντα 2020 και πιστεύουμε ότι πρέπει να εστιαστούμε ιδιαίτερα ε, στην ε, ενίσχυση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, στην αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών για την ασφάλεια και το περιβάλλον, την ενίσχυση της θέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίω όσον αφορά την έρευνα και την τεχνολογία. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να υπάρχει συμπληρωματικότητα και συνεργασία ε, στο θέμα της χρηματοδότησης για την ε, ε, έρευνα και την ανάπτυξη μέσω της πολιτικής συνοχής, της κοινή γεωργικής πολιτικής και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση και άλλα, και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Συμφωνούμε ότι το πρόγραμμα Horizon 2020 πρέπει λογικά να μειώσει τον κατακαιρματισμό και να αυξήσει τη συνοχή συμπεριλαμβανομένων των εθνικών προγραμμάτων έρευνας ο συντονισμός της έρευνας και της ε, καινοτομίας είναι προτεραιότητα για την, Ευρωπα... για την Δανική Προεδρία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, θέλουμε να υπάρχει επιλεκτική χρηματοδότηση για τα ε, προγράμματα ε, καινοτομία και θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια ισχυρή ανεξάρτητη Ευρώπη της καινοτομία. Επίσης, το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να ενισχύσει την ευελιξία στο πρόγραμμα πλαίσιο, κάτι που είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προϋπόθεση για, να, για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και ευνοεί ιδιαίτερως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λιγότερη γραφειοκρατία εργασία, περισσότερη έρευνα, αυτό θα είναι η εποδός μας. Θα ήθελα να πω τώρα μερικά πράγματα για το πώς ε, ε, θα λειτουργήσει η Προεδρία μας. Ε, είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον ορίζοντα 2020. Το χρονοδιάγραμμα είναι δύσκολο αν θέλουμε το νέο πρόγραμμα να είναι έτοιμο το 2014. Συνεπώς πρέπει να ε, θέσουμε έναν φιλόδοξο στόχο. Ο στόχος μας είναι οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν ε, όσο το δυνατόν συντομότερα στο πλαίσιο της Προεδρίας μας. Θα θέλαμε δηλαδή να ε, φτάσουμε σε μια γενική προσέγγιση για τον ορίζοντα 2020 στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού στις 31 Μαρτίου του 2012. Στην πρώτη φάση της ε, Προεδρίας μας ε, θα συζητήσουμε τις διάφορες απόψεις για τον ορίζοντα 2020 με τους βασικούς εμπλεκομένους φορείς ε, της Ευρώπης. Έχουμε μια υπουργική διάσκεψη στην Κοπενχάγη 21 Φεβρουαρίου 2012 για το διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς για τον ορίζοντα 2020 η υπουργική διάσκεψη είναι ακριβώς πριν από τις 2 Φεβρουαρίου που θα γίνει μια ανεπίσημη συζήτηση σε υπουργικό επίπεδο για τον ορίζοντα 2020 και χαιρετίζουμε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτά τα ε, σε αυτές τις ε, ε, συζητήσεις και έχουμε καλέσει και την βασική εισηγήτρια για να συμμετέχει. Στις 21 Φεβρουαρίου θα γίνει μια συζήτηση προς ανατολισμού για τον ορίζοντα 2020 Επίσης έχουμε προβλέψει ένα ανεπίσημο σεμινάριο το Μάρτιο ή τον Απρίλιο να γίνει εδώ μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα οργανωθεί από κοινού με την, ε, από τη Δανική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μια ανεπίσημη συζήτηση ε, κατά την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων για τον ορίζοντα 2020. Και είμαι ε, πεπισμένος ότι το σεμινάριο αυτό θα, θα συνεισφέρει σημαντικά στις ε, επερχόμενες συζητήσεις. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η Προεδρία μας θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να εξασφαλίσει την βέλτιστη δυνατή ε, συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συνεργασία μεταξύ των θεσμών, με τους ερευνητές, ε, με τη βιομηχανία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, ένα σημαντικό στοιχείο για την ε, ε, βελτίωση ε, της ανταγωνιστικότητάς μας και θα γίνουν πολλές συζητήσεις και με την Κύπρο και την Πολωνία. Νομίζω ότι αν καταφέρουμε να, κατα... να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς θα, γεφυρά... θα γεφυρώσουμε οποιαδήποτε χάσμα υπάρχει μεταξύ του προγράμματος πλαισίου και του προγράμματος ορίζοντα 2020. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και είμαι διαθέσιμος για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Στεργκάρντ, ο οποίος ε, σεβάστηκε και το χρόνο του, τον οποίο του διαθέσαμε. Τον ευχαριστούμε θερμά και τώρα δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να εγγραφεί στο κατάλογο των ομιλητών. Ε, να ξεκινήσουμε με την κυρία Δελκαστήγιο για να ξεκινήσουν οι αγορητές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είναι αξιοζήλευτη η Προεδρία σας για κάθε κράτος μέλος που έχει αναλάβει την Προεδρία. Το θέμα της ενεργειακής απόδοσης θα σας απασχολήσει αυτό το διάστημα και επίσης και ένα από τα προγράμματα τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή κοινοτική χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα για την έρευνα στο πακέτο Horizon 2020. Εδώ στο Κοινοβούλιο λοιπόν και στην Επιτροπή μας πιο συγκεκριμένα, πραγματικά θα βρεθείτε ενώπιον πάρα πολλών μελών, όπως βλέπετε, που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και για τη μία και για την άλλη πτυχή και νομίζω ότι έχουν και πολύ υψηλέ ε, δεξιότητες και πυρογνωμοσύνη επί του ζητήματος, κάτι το οποίο φυσικά είναι πολλά υποσχόμενο. Θα ήθελα να σας επισημάνω κάποιες πτυχές, οι οποίες κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα σημαντικές ε, ε, δεν είναι όλες βέβαια, είναι κάποιες, έχω σταχυολογήσει κάποια στοιχεία διότι θα έχετε πολύ, χρόνο, ε, πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή σας και εσείς ξέρετε τι γίνεται με τα χρονικά όρια στις επιτροπές, αλλά επειδή μέχρι τούδε η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πάρα πολύ καλή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχθηκε πολλές από τις προτάσεις που έγιναν από πλευράς Επιτροπής μας ώστε να ετοιμάσουν τελικώς το έγγραφο που μας παρουσίασαν, υπάρχουν όμως ακόμα πολλές ε, δυνατότητες βελτίωσης. Και ακριβώς αυτές οι δυνατότητες βελτίωσης είναι αυτές στις οποίες θα επικεντρωθεί η Επιτροπή μας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας αναφέρω τρεις επιγραμματικά. Το ένα είναι το γενικό θέμα της χρηματοδότησης. Ανησυχούμε ιδιαίτερα διότι η χρηματοδότηση λογικά ε, καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις προτεραιότητες που θα καθοριστούν. Εάν δεν συμβαδίζουμε εκ παραλίλου δεν μπορούμε να εγκρίνουμε κάποια στοιχεία χωρίς να γνωρίζουμε αν θα υπάρξει και αντίστοιχη στήριξη μέσω προπολογισμού. Και δεν θα έχουν και καμία αξία. Εάν ξέρουμε πώς θα πάει η χρηματοδότηση, μπορούμε να καθορίσουμε προτεραιότητες μεταξύ των στόχων που θεωρούμε ότι είναι οι πιο ενδιαφέροντες. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο ε, σημείο είναι στην ουσία δύο πράγματα τα οποία θα ήθελα να φέρω. Το ένα το γνωρίζουμε ως τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Εδώ υπάρχει ένα πλεονέκτημα γιατί δεν έχουμε πολλές καινοτομίε ε, σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθούν πολύ περισσότερα κίνητρα για τα μέσα ώστε να υπάρχει ένα πραγματικό άνοιγμα των εθνικών προγραμμάτων. Διότι υπό μία έννοια με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε το κέντρο της Ευρωπαϊκής ε- Έρευνας, το ERA. Και αυτό δεν είναι πολύ σαφές. Ε, εδώ, στη δέσμη των μέσων, πρέπει να δοθούν προτεραιότητα σε προγράμματα ή δράσεις, που μπορεί να είναι και μικρά προγράμματα ή μικρές δράσεις, διότι θα δώσουν το έναυσμα για μεγαλύτερα προγράμματα και έτσι μπορεί να προκύψουν και προγράμματα από μικρές επιχειρήσεις και από πανεπιστήμια. Ε, σκεφτόμαστε συνέχεια τα μεγάλα προγράμματα αλλά δυστυχώς ε, ε, παραλείπουμε τα μικρά και αυτό είναι σημαντικό. Και τέλος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας το Κοινοβούλιο, υπήρχε και μια έκθεση στην οποία ήταν ε, η συγχύτρια συνάδελφος ε, Καρβάλιο και συνεισέφερε ιδιαίτερα στο θέμα της απλούστευσης, που πάντα ήταν η μεγάλη εκκρεμότητα, αν θέλετε, στα προγράμματα πλαίσιο. Ακόμα και έτσι όμως υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία θα μπορούσαμε να τελειοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω λοιπόν κάποιες πτυχές. Μία πιο συγκεκριμένα. Ίσως θα ήταν καλή στιγμή για να αυξηθεί δραστικά η πληρωμή ε, για το ότι υλοποιήθηκε μέσα στις κοινοπραξίες και δεν έγινε. Και θα πρέπει να την αξιολογήσουμε αυτή την πτυχή. Είναι κάτι το οποίο θα μείωνε πολύ σημαντικά το κόστος διαχείρισης των προγραμμάτων και είναι αυτό το οποίο επιθυμούν όλοι στον τομέα της έρευνας. Αυτό ήλπιζαν. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Δόθηκε ένα σημαντικό βήμα ε, σε θέματα απλούστευσης και έτσι υπάρχει χώρος διαθέσιμος για να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, εμείς δεσμευόμαστε ε, να συνεργαστούμε μαζί σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ντελκαστήγιο και τώρα ο λόγος στην κυρία Ριέρα Μαντουρέλ, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εξ ονόματο τη ομάδα μου, σα καλωσορίζω εδώ στην Επιτροπή μα και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για όλε τι εξηγήσει που μα δώσατε ε, και να σα πω εκ των προτέρων ότι συμφωνώ με την πλειοψηφία των ε, θεμάτων που έχετε στο πρόγραμμά σα για την Προεδρία σα, ε, στην οποία έχουμε αναποθέσει πάρα πολλέ ελπίδε. Όπω είπε και η κυρία Ντελκαστήγιο, είναι κλειδί η χρονική συγκυρία για την καινοτομία και την τεχνολογία και την έρευνα. Ξεκινάει η συζήτηση την εφαρμογή του νέου προγράμματος πλαίσιο Horizon 2020 ε, και παρά το γεγονός ότι θα εγκριθεί την επόμενη χρονιά, ο προσανατολισμός που θα του δοθεί από την πρώτη στιγμή είναι κλειδί και επομένως για τους επόμενους μήνες ε, θα έχουμε πολύ σημαντική δουλειά και θα είναι πολύ σημαντικοί αυτοί οι μήνες προς αυτή την κατεύθυνση και εσείς μπορείτε να συνεισφέρετε ιδιαίτερα στους τομείς αυτές, ιδίω στον τομέα της καινοτομίας όπου η πείρα σας είναι αναγνωρισμένη από όλους. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Συμφωνώ, όπως σας είπα και με τα περισσότερα από όσα μας είπατε και χωρίς να επαναλαμβάνω τα όσα είπε η κυρία Αντελκαστήγιο προηγουμένως, θα ήθελα και εγώ να επικεντρωθώ σε μία-δύο πολύ συγκεκριμένε πτυχές της πρότασης που μας έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Horizon 2020. Πρόκειται για πτυχές που διαβάζοντας τα έγγραφα τα οποία μας έδωσε η Προεδρία, Φαίνεται ότι έχουν υπογραμμιστεί ε, στις θέσεις που είχαμε από πέρσι και θα ήθελα να τις προασπίσετε κι εσείς κύριε Υπουργέ ως Προεδρία διότι η ομάδα μας πραγματικά θα ήθελε να συμπεριληφθούν στην τελική μας θέση. Το πρώτο είναι το θέμα της απλούστευσης. Η κυρία Δελκαστήγιο σας έδωσε παραδείγματα. Το Υπουργείο σας ζητούσε εκβάθρον απλούστευση ε, βάσει των πληροφοριών που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας και εμείς... Ε, ε, κατανοούμε μεν ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά και ίσως δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει, αλλά ε, θεωρώ ότι η πρόταση που μας έκανε δεν ικανοποιεί στο 100% το στόχο της απλούστευσης. Θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι και όπως σας έλεγα, λαμβάνοντας υπόψη ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι το ζήτημα αυτό και τι δυσκολίε συμπεριλαμβάνει, θα θέλαμε να προχωρήσουμε περαιτέρω το ζήτημα αυτό και βασιζόμαστε στην υποστήριξή σας και θα θέλαμε να ξέρουμε και την άποψή σας επί του ζητήματος. Μια άλλη προτεραιότητα είναι οι υποτροφίες Marie Curie. Τις αναφέρατε κι εσείς και εμείς συμφωνούμε και δεχόμαστε ότι είναι αναπόσπαστο τμήμα ε, για τους νέους ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν την επιστημονική τους καριέρα στην Ευρώπη και είναι και φυσικά ε, στοιχείο της ανταγωνιστικότητάς μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο προπολογισμός δεν είναι ο κατάλληλος για αυτές τις δράσεις, δεν ξέρω τι άποψη έχετε εσείς και δεν θεωρούμε ότι αναπτύχθηκε κάτι σημαντικό που είναι το γεφύρωμα με τη βιομηχανία που αναφέρατε κι εσείς. Θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα στο οποίο θα μπορούσαμε να πάμε έτσι περαιτέρω και θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Και τέλος, τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, εσείς λέτε ότι ε, περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, αλλά θα θέλαμε να μας απαντήσετε στο εξή. Θεωρείτε ότι ίσως θα ήταν καλύτερα αφού συμφωνήσουμε σε ένα περιορισμένο αριθμό προκλήσεων να καθορίσουμε έναν ορισμό βάσει τον οποίο θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε περισσότερα προγράμματα σε κάθε μία από αυτές τις πτυχές. Μήπως ε, ο περιορισμός αυτός θα πλήξει και τον αριθμό των πιθανών προγραμμάτων που θα εγκρίνουμε. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και θα θέλαμε να αναφέρουμε ευθύ εξ αρχής. Να σας πω επίσης ότι όλα όσα είπατε, το να υπάρχει μερική συμφωνία στο τέλος της Προεδρίας σας για τα βασικά ζητήματα είναι πολύ καλή ιδέα. Ό,τι μπορούμε να προχωρήσουμε από πλευρά συμφωνιών είναι σημαντικό και επίσης ως εισηγήτρια του Horizon 2020 η επιθυμία μου ε, είναι να συνεργαστούμε εξ αρχής με όλους τους και εισηγητές αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο αυτή εξ αρχής ώστε να καταφέρουμε να έχουμε σημαντικές συμφωνίες ε, που είναι και τόσο σημαντικές για το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλους συντονιστές εγγεγραμμένους και έχουμε 10 ακόμα παρεμβάσεις. Κλείνει ο κατάλογος των αγορητών, τρία λεπτά ο καθένας ε, για να μπορέσουν να λάβουν το λόγο όλοι και να ακούσουμε και τον Υπουργό. Ο κύριος Βάλτσιτς. Ε, Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, όντως η η μερίσια διάταξη της Δανειγικής Προεδρίας είναι πολύ φιλόδοξη και μπορούμε απλώς να συγχαρούμε τη Δανία που σε αυτή την περίοδο κρίσης ε, καταφέρνει να εφαρμόσει το φιλόδοξο πρόγραμμά της. Έχω μία ερώτηση όμως. Η στρατηγική για το 2020 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προβλέπει ε, πολλές ανησυχητικές προοπτικές δημογραφικά παραδείγματος χάρη και θα πρέπει όλοι καθώς και η Δανία να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα της υγειονομικής περιθάρψεως. Θα φροντίσετε λοιπόν να υπάρξει κάποια μνήμα ε, για τα θέματα της ε, κοινωνικής και υγειονομικής προστασίας διότι αυτός ο τομέας είναι καινοτόμος και για πολλούς για μας θα είναι πολύ περίπλοκο να το κατανοήσουμε. Εσείς λοιπόν κύριε Υπουργέ θα ήθελα να μας παρουσιάσετε ορισμένα σχόλια επί του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Τζόνσον. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω ότι ε, ο Ιδανός Πρόεδρος έθεσε το, αυτό το θέμα τόσο καλά διότι και εγώ είχα συμμετάσχει σε μία συνάντηση της Δανικής Προεδρίας με την Επιτροπή μας και ε, όντως ε, διαπίστωσα ότι είχε εξαιρετικά εισάγει το θέμα. Επί πλέον έχω την εντύπωση ότι οι εκπρόσωποι του Δανικού Κοινοβουλίου συνεργάζονται πάρα πολύ στενά και καλά με την Προεδρία και πρέπει να σας πω ότι ενώματι της πολιτικής μου ομάδας θα είμαι εκπρόσωπος και θα συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα Horizon 2020 που είναι κάτι που με χαροποιεί πολύ. Πλέον αυτού, σαν εκπρόσωπος της ομάδος των φιλελευθέρων, θέλω να αναφερθώ εις, ε, εις ε, εργασίες για την καινοτομία στο σκανδιναβικό χώρο που όπως τόνισε και ο, ο κύριος Υπουργός είναι ένας ε, τομέας προτεραιότητος και ε, θα δραστηριοποιηθούμε από την αρχή. Θέλω όμως πέραν αυτού να κάνω δύο ερωτήσεις. Αφενός ε, θα θέλαμε να ενισχύσουμε το input, δηλαδή πρέπει να ενισχύσουμε το input αλλά από την άλλη πλευρά όλα αυτά θα πρέπει να λειτουργούν εύρυθμα διότι πολλές φορές οικονομικά ε, επενδύουμε πολλά αλλά ε, τα αποτελέσματα ε, δεν είναι ικανοποιητικά οπότε και αυτά θα πρέπει να στηριχθούν. Και εδώ συμφωνώ με αυτούς οι οποίοι είπαν ότι χρειαζόμαστε μεν τα μέτρα αλλά θα πρέπει να λειτουργούν και σωστά. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι από τη μία πλευρά έχουμε σημαντικές ε, ε, ε, επενδύσεις αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται από μείωση της γραφειοκρατίας ώστε να επιτρέψουν και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στα μικρότερα ερευνητικά προγράμματα. Δεύτερον, χρειαζόμαστε μία σειρά μέτρων κατά τρόπον ώστε ε, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με εκπροσώπους πορών κρατών μελών σε περιφερειακό επίπεδο οποίο θα πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά και θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε διάφορους τομείς. Αυτό θα μπορεί να περιληφθεί στην ε, στρατηγική για το 2020 και να συνδυαστεί με την πολιτική συνοχής. Εδώ πρόκειται ε, επίσης ε, για τον τομέα της αριστείας στον ορίζοντα 2020 και στη βελτίωση της υποδομής. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αναπτυχθεί για να καταλήξουμε σε αριστεία. Ακριβώς αυτή η αριστεία θα πρέπει να εφαρμοστεί ευρέως σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και τέλος πιστεύω ότι εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχουμε ενεργά στο πρόγραμμα Horizon 2020 να, να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και ελπίζουμε ότι οι εκπρόσωποι των διαφόρων κρατών μελών θα συμβάλλουν κατά τρόπον ώστε να παραμείνουμε ε, εστιασμένοι και ε, συσπηρωμένοι ε, προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία η οποία είναι πολύ σημαντική και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι να προωθήσουμε την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ. Ε, χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για την ε, επίσκεψη αυτή της Δανικής Προεδρίας στην Επιτροπή μας διότι ε, εδώ ξεκινήσαμε ήδη την εργασία στον τομέα του ορίζοντα για το 2020 ίσως δεν ολοκληρώσει το έργο η Προεδρία αλλά έχει παρουσίασει πλησιάσει καλά την αρχή. Ε, Χθε ήρθε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μας παρουσίασε το πρόγραμμα Horizon 2020 και ελπίζουμε ότι θα πρέπει ε, να προχωρήσουμε από τις θεματικές ενότητες αυτού του προγράμματος σε ε, νέα θέματα διότι αυτά που μας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως είναι ο τομέας του κλίματος και της υγείας και την περασμένη εβδομάδα το Πανεπιστήμιο της Κοπεχάγης έκανε μία θαυμάσια παρουσίαση στις Βρυξέλλες για το θέμα της καταπολεμήσεως της ασθενείας του διαβήτη και τα παρουσίασαν, παρουσίασαν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Χαίρομαι για αυτές τις εξελίσεις αλλά έχω παρόλα αυτά και ανησυχίες. Είμαι ε, κοινωνική λειτουργός και βλέπω ότι ορισμένες πτυχές δεν περιλαμβάνονται πια στο πρόγραμμα και ε, βλέπουμε ότι παραμένει μένει ατομική φυσική χωρίς όμως να βλέπουμε άλλα, άλλους σημαντικούς τομείς υπάρχουν μεγάλες επενδύσεις και ε, στην Επιτροπή μας έχουμε ένα ερευνητικό συμβούλιο για να να υπάρξει έρευνα σε όλους τους τομείς και να λαμβάνονται αποφάσεις τεκμηριωμένα όχι σαν να ήμασταν ένας α, ε, γενικός ιατρός. Άρα οι κοινωνικές επιστήμες θα πρέπει και αυτές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και βλέπω ότι εδώ δεν προβλέπεται καμία επένδυση για τον τομέα αυτό. Ε, δεν προβλέπουμε επενδύσεις για την έρευνα στον τομέα της οργανωμένης εγκληματικότητας των κλιματολογικών αλλαγών και εάν διάφορες πτυχές δεν εξεταστούν θα πρέπει να βρεθούν διαφορετικοί πόροι για έρευνα στον τομέα αυτό και διαπιστώνω ότι στο London School of Economics εξετάζουν πώς θα αντεπεξέλθουμε τις κρίσεις και θα έπρεπε και η ιδανική προεδρία να ταχθεί κατά τρόπον ώστε να προχωρήσουμε στον τομέα των κοινωνικών επιστημών και ε, ε, άλλο. Η κυρία Χέρτσοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ την Πρόεδρό μας για την εκλογή της, στη θέση της Προεδρίας. Δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνω χθε ε, και θα ήθελα να κάνω και μερικές ερωτήσεις ε, στον Υπουργό. Χρειαζόμαστε τον αθλητισμό. Χρειάστηκε να κάνουμε οικονομίες αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω να αναφέρεστε περισσότερο σε καινοτομία, περισσότερο στον αθλητισμό, πώς θα μπορέσουμε να ε, εξασφαλίσουμε ότι τα καλά μυαλά δεν θα φεύγουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ότι οι πόροι θα παραμένουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε χωρίς να ε, χρειαστεί να δαπανίσουμε μεγαλύτερα ποσά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί. Έχω τρεις μικρές ή μεγάλες ανησυχίες. Καταρχήν μας είπατε ότι η έρευνα στον τομέα τον επιστημονικό είναι σημαντική για μας, ιδίω τονίσατε στις πράσινες επιστήμες. Θα ήθελα να διευκρινίσετε παρακαλώ, διότι το μέλλον της Ευρώπης δεν είναι μόνο στις πράσινες επιστήμες αλλά και στις παραδοσιακές επιστήμες διότι ορισμένες χώρες άντεξαν καλύτερα στην κρίση διότι προωθούσαν τις παραδοσιακές βιομηχανίες, χαλιβουργία, χημική βιομηχανία, βιομηχανία οπότε θα πρέπει και στις παραδοσιακές αυτές βιομηχανίες να επενδύσουμε στο μέλλον. Επίσης ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένως είναι ότι ορισμένα κράτη δεν έχουν συμμετάσχει στην έρευνα σε μεγάλα θέματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι όλοι συμφωνήσαμε ότι η αριστεία είναι σημαντικό θέμα αλλά δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε με ένα ποτιστήρι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός μεταξύ ε, κρατών που είναι ε, πιο ε, προχωρημένα στην έρευνα και να υπάρχει μία άμυλα με χώρες οι οποίες δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες στον τομέα της έρευνας για να υπάρχει και ανάπτυξη και ενίσχυση αλλά και πρόοδο στην έρευνα. Εάν δεν έχουμε περισσότερους πόρους διαθέσιμους, το οποίο μπορεί επίσης να συμβεί και πρέπει να επιβιώσουμε με συρρυκνωμένους πόρους, το οποίο να πέφχομαι, θα έπρεπε να έχουμε βασικά θέματα και να αξιολογήσουμε τι είναι πιο σημαντικό και τι πιο επουσιώδες. Και αυτή, η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνει διαρθρωτικά για να μην τσακωνόμαστε μεταξύ κρατών διότι ίσως καλό θα ήταν να μας δώσετε κάποια ένδειξη του πώς κλείνει η πλάστιγκα στον τομέα αυτό. Ο κύριος Βέμπερ. Θα ήθελα και εγώ να ε, σας συγχαρώ Συμφωνούμε με τη φιλοδοξία την οποία, στην οποία αναφερθήκατε, τη συμμεριζόμαστε. Αν θα έπρεπε να τα ξανακάνουμε όλα από την αρχή, εγώ θα ξεκινούσα από τον πολιτισμό. Ουσιαστικά αρχίσαμε όμως από τον άνθρακα και το χάλιβα. Ο άνθρακας και ο χάλιβας του 21ου αιώνα όμως είναι η έρευνα και η καινοτομία. Έχετε λοιπόν ε, ένα καθοριστική σημασία χαρτοφυλάκιο να λάβει και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει όλο και μεγαλύτερη καθυστέρηση σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να ε, συζητήσουμε το θέμα υπό μία λίγο δύο διαφορετική οπτική γωνία. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη του, της έρευνας και της καινοτομίας είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα λαιλασίας των ε, πόρων αυτών. Η πνευματική ιδιοκτησία συνεχώς παραβιάζεται και όχι μόνο από την Κίνα, πώς έχετε σκοπό να υπερασπιστείτε τις ευρεσιτεχνίες μας, την τεχνολογία μας, τη δική μας ε, ε, ε, ιδιοκτησία, την πολιτιστική και την πνευματική, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο γίνεται όλο και περισσότερο επίγον. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να επενέσω τον ε, Υπουργό για την ε, παρουσίασή του και κυρίως τη σαφήνεια των στόχων και, της αποφασιστικό, την αποφασιστικότητά του για τους επόμενους έξι μήνες ε, και επειδή εγώ μόλις έρχομαι από την συνεδρίαση της, της Επιτροπής Πολιτισμού όπου άκουσα και εκεί συναδελφό σα, είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι υπάρχει πλήρης συνεργασία και συντονισμός το Εράσμους, η έρευνα, η καινοτομία κλπ. Αναφερθήκατε στη ε, σημασία της ολοκλήρωσης της ενιαίας ε, αγοράς. Τι μπορείτε να κάνετε εντός έξι μηνών για να προσπαθήσετε να το καταφέρετε αυτό και δεδομένης ε, της, του, ιστορικού, της, δεδομένου του ιστορικού της χώρας σας για, στην πράσινη οικονομία προγράμματα ή πρωτοβουλίες για βέλτιστες πρακτικές οι οποίες πρέπει να γνωστοποιηθούν στο ευρύτερο κοινό ε, έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο ώστε να μπορέσουμε και εμείς να επιτύχουμε ευκολότερα τους στόχους μας για το 2020. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τζόνταν Τζιζέλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τις ε, σαφέστατες παρουσιάσεις σας, για τις προτεραιότητες ε, της Προεδρίας σας. Θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο ορίζον 2020 γιατί είναι τόσο σημαντικό, πρέπει να έχουμε κατά νου και τις αποφάσεις οι οποίες λήφθησαν σε υπουργικό επίπεδο και ε, να αναλάβουμε και δράση για να υλοποιηθούν αυτές. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνες. Ξέρετε ότι εδώ βαδίζουμε με βήματα χελώνας. Θα μας βοηθήσουν όμως ε, τα βήματα αυτά να ε, υλοποιήσουμε τα αποτελέσματα και των προγράμματων πλαίσιο. Υπάρχει ε, η απόφαση για τη λεγόμενη πέμπτη ελευθερία, για την ελευθερία μετακίνησης της επιστήμης στη Λουμπλιάνα. Τι ε, σχέδια έχετε για περαιτέρω έρευνα για την εναρμόνιση των κρατών μελών στις ερευνητικές τους πολιτικές. Τι προγράμματα, τι σχέδια έχετε συγγνώμη, για τις συνέργειες και τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι υπουργοί στις χώρες τους ταυτόχρονα με τις αποφάσεις για το ορίζον 2020. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φανλίστερ, Λόραϊ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να προσθέσω κάποια πράγματα. Καταρχάς να σας πω ότι ανησυχώ. Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την κατάστασή μας κατά 30-40% περισσότερο, θα υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία θα θέλουν πάντα να μειώσουν το ποσοστό της συνεισφοράς τους. Εσείς είστε προεδρεύον του Συμβουλίου. Πώς ε, διαχειρίζεστε την όλη διαδικασία μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα προς το μέλλον ή θα σταματήσουμε, θα μείνουμε στάσιμοι. Πώς ε, βλέπετε το θέμα ε, και από την πλευρά του διεθνούς προϋπολογισμού. Δεύτερη ερώτηση. Τι κάνετε με τις μεγάλες επενδύσεις οι οποίες πρέπει να έχουμε για τις ε, υποδομές έρευνας. Υπάρχουν κάποιες επενδύσεις ε, που γίνονται σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης, αλλά όχι παντού. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, δεν μας επιτρέπεται αυτή η πολυτέλεια. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν τα θέματα αυτά. Και τέλος, εν κατακλείδη, αναφερθήκατε στις ε, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό το οποίο ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το γεγονός ότι εσείς στη Δανία έχετε πολύ καλή πείρα επί του θέματος. Από τεχνολογική σκοπιάς μπορούμε να έχουμε μια κάποια πρόοδο, αλλά ε, επειδή ε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την Κίνα, σταματούν όλα. Τι θα γίνει, πρέπει να λάβουμε υπόψη του διάφορου τομεί. Παραδείγματο χάρη, ηλιακή ενέργεια. Πώ θα το αποφάσουμε, πώ μπορούμε να το υλοποιήσουμε, πώ μπορούμε να εξετάσουμε τα θέματα αυτά. Και τέλο, όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μα για να έχουμε περισσότερους πόρους. Το Risk Sharing Facility υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. με 2 δισεκατομμύρια συνεισφορά, ε, καταφέραμε να έχουμε επενδύσει 16 δισεκατομμυρίων. Πώς θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ κυρία Τόγια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, καταρχά να συγχαρώ και εγώ τη Δανική Προεδρία και εσά, κύριε Υπουργέ για τη σαφήνεια και τη φιλοδοξία των προτάσεών σας. Ε, Σημερίζομαι και εγώ το χρονοδιάγραμμα που προτείνατε και αυτή την κοινή πρωτοβουλία μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για να ε, διοργανώσουμε ένα εργαστήριο, ένα συνέδριο εδώ στο Κοινοβούλιο για να ενισχύσουμε την ε, διοργανική μας συνεργασία. να προσθέσω κι εγώ κάποια στοιχεία συμφωνώντας με τις περισσότερες παρεμβάσεις της κυρίας Μαντουρέλ και των υπορρήπων. Περιμένουμε πολλά από την Προεδρία σας, ε, αυτό το μεγάλο κεφάλαιο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Πού θα καταλήξουν, θα γίνουν ένας τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα υπόλοιπα προβλήματα, θα ενσωματωθούν παντού και θα γίνουν αναπόσπαστο σημείο όλων ή θα εξαφανιστούν ως κάτι πολύ εξειδικευμένο και θα χάσουν την αξία τους. Εμείς ε, θεωρούμε ότι το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί ε, να επιτρέψει στον εαυτό του να χάσει αυτή τη σημαντική πτυχή. υπάρχει ε, και στη χώρα σας ε, πολύ μεγάλη πρόοδο σε κοινωνική καινοτομία, τις υπηρεσίες, ε, αναφερθήκαμε και στην πνευματική υγεία. Υπάρχουν όλες αυτές οι προκλήσεις λοιπόν για το μέλλον και περιμένουμε πάρα πολλά από την εμπειρία της Δανίας και τη συνεισφορά της. Μας ενδιαφέρει επίσης και το πώς η έρευνά μας μπορέσει να αποτελέσει προγεφύρεμα για την ε, βιομηχανική ανάπτυξη. Το αναφέραμε και στο θέμα που προηγήθηκε της άφηξής σας και θα ήθελα να αναφέρω αυτό που είπε και ο κύριος Βέμπερ. Πώς μπορούμε να καταφέρουμε όλος ο προγραμματισμός που γίνεται, ο οποίος με το πρόγραμμα πλαίσιο αυξάνεται, να γίνει και ικανότητα των βιομηχανιών μας, να γίνει προϊόν, να υλοποιηθεί σε κάτι, να είναι κάτι χειροπιαστό στην Ευρώπη. Εχθές ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ρωτήθηκε από πλευράς μου τι έγιναν ε, διάφορες, ε, διάφορα πορίσματα ομάδων υψηλού επίπεδου και η απάντηση ήταν ότι έγινε δεκτό μέσω του Deploy in Europe First. Μπορούμε να έχουμε κάτι από αυτή την πτυχή. Τα προγράμματα τα οποία επιλέγουμε και από τη συμφορά μας στην Ευρωπαϊκή Έρευνα μπορούμε να τα προωθήσουμε και λίγο περισσότερο ώστε να γίνουν προγράμματα τα οποία θα μεταφραστούν σε προϊόντα στην Ευρώπη χωρίς να γίνουμε προστατευτικοί. Αλλά το θέμα της ε, ε, προστασίας των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για παράδειγμα και πώς μπορεί να γίνει ένα προϊόν που θα γίνεται εδώ στην Ευρώπη. Ίσως το Deploy in Europe First να είναι λίγο υπερβολικό αλλά το να μας ενδιαφέρει ε, και το ε, πώς υλοποιούνται τα αποτελέσματα της έρευνας πάλι είναι λίγο. Πού μπορούμε να βρούμε τη χρυσή τομή σε αυτά. Ευχαριστώ κύριος Πρόντι. πολύ σύντομα, διότι τα περισσότερα θέματα αναφέρθηκαν επανειλημμένως. Θα ήθελα να σταθώ και να υπογραμμίσω την ανάγκη μεγαλύτερης κινητικότητας των ερευνητών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διευκολύνουμε αυτές τις αλλαγές, τις ανταλλαγές σε όλους τους τομείς που αναφέρθηκαν και που είναι πολύ σημαντικοί για το μέλλον της Ευρώπης. Αναφέρομαι για παράδειγμα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τον οδικό χάρτη για την Ευρώπη χωρίς άνθρακα για το 2050. Πρόκειται για μια τεράστια διαδικασία η οποία θα πρέπει να ε, εξεταστεί και λίγο πιο συγκεκριμένα ως προς την οργάνωσή της και την υλοποίησή της, διότι είναι μία πρόκληση που είναι ανάλογη αυτού που χαρακτήρισε δυστυχώς την Ευρώπη και τον κόσμο μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, είναι δηλαδή θέματα τα οποία κατά την άποψή μου θα πρέπει να τα σκεφτούμε λίγο καλύτερα από συστημική σκοπιά και να ξεκινούμε από την ανάγκη της ε, ισχυρής ανάπτυξης και της έρευνας, η οποία θα είναι αυτή που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ε, τελευταίος ο κύριος Ρόντε και μετά θα λάβει το λόγο ο Υπουργός. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να ζητήσω το λόγο γιατί έχουμε και άλλες ε, ε, ευκαιρίες να συζητήσουμε αλλά υπάρχει κάτι το οποίο με ενέπνευσε πάρα πολύ ο κύριος Ρόιλ μίλησε πριν από μένα και αυτός αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα δηλαδή είπα σχέτως αν έχουμε περισσότερη χρηματοδότηση ή όχι θα πρέπει να είμαστε τολμηροί να καταρτήσουμε μία, έναν κατάλογο προτεραιοτήτων και αυτό είναι σημαντικό μία κατάρτιση προτεραιοτήτων δυστυχώς όμως το τότε θα υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι πιστεύουν ότι ε, πρέπει να διαλέξουμε τους ε, νικητές, pick the winners. Οπότε θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη της ε, Δανικής Προεδρίας. Διαλέγουμε μόνο τους νικητές, δηλαδή αυτούς που είναι στην συμπολίτευση. Αυτό πιστεύουν ορισμένοι και θα ήθελα εδώ να σας προειδοποιήσω. Είναι πολύ δύσκολο για τους πολιτικούς να προεξοφλήσουν ποιος θα κερδίσει στο μέλλον και θα πρέπει καταρχήν να καταρτήσουμε ένα σωστό πλαίσιο, να αφήσουμε τους ερευνητές να δουλέψουν και να μην προεπιλέγουμε τους νικητές, να μην δηλαδή εξασκήσουμε μία στρατηγική pick the winners. Ευχαριστώ. Ήσασταν όλοι πολύ καλοί, σεβαστήκατε τα χρονικά περιθώρια, επομένω μπορούμε να δώσουμε 10 λεπτά με ηρεμία στον Υπουργό να απαντήσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για τις πολλές ερωτήσεις. Ε, κάτι το οποίο δείχνει πραγματικά ιδιαίτερη αφοσίωση από πλευράς της Επιτροπής σας, ε, τουλάχιστον για τις διαπραγματεύσεις για τον ορίζοντα 2020 και την ανάπτυξη ε, μια ναι, την ανάπτυξη του μεγαλύτερου και πιο πλούσιου προγράμματος ερευνητικού στον κόσμο. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν με την ε, κυρία Τελκαστήλιο που είπε ότι υπάρχει περιθώριο βελτιώσεως βεβαίως ε, και ελπίζω ότι αυτό θα καταφέρουν οι διαπραγματεύσεις. Θα μπορέσουμε δηλαδή να βελτιώσουμε όπου πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Αναφερθήκατε σε τόσο πολλά ζητήματα, θα προσπαθήσω κάπως να τα ομαδοποιήσω. Πρώτον, θα ήθελα να αναφερθώ στην απλοποίηση. Νομίζω ότι όλοι είναι υπέρ της απλοποίησης, ε, κανένας... Ε, ε, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά χωρίς να μας ρωτάει κάποιος ή να επιμένει κανείς για την απλοποίηση. Και, απλοποίηση. και επειδή βέβαια ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, να μην σας πω στον αριθμό των λεπτομεριών, θα ενθαρρύνω τους συναδέλφους όταν θα γίνει η ανεπίσημη συνάντηση στην Κοπενχάγη την επόμενη εβδομάδα να υποβάλουμε προτάσεις οι οποίες θα απλοποιούν και όταν θα συνεχίσουμε ε, τη δουλειά μας, όχι μόνο στην αρχή των διαπραγματεύσεων αλλά και στο τέλος, ε, να θυμόμαστε πάντοτε την ε, δέσμευσή μας για την απλοποίηση, ειδικότερα όσον αφορά συγκεκριμένες τροποποιήσεις όταν θα φτάσουμε τέλος πάντων στην, στο, στην τελική πινελιά να το έχουμε υπόψη μας. Νομίζω ότι η απλοποίηση είναι ένα απαραίτητο βήμα για να μπορέσουμε να ε, καταφέρουμε κάτι το οποίο αναφέρατε πολύ, δηλαδή την ε, δυνατότητα, της, τη δυνατότητα συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή ε, μικρότερων κοινοπραξιών. ο κύριος Γιώχανσον αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα και ο αριθμός των ερωτήσεων γενικώ για την απλοποίηση δείχνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάει επιτέλους μπροστά αυτό το ε, θέμα. Το Κοινοβούλιο και η δική σας Επιτροπή έχει κάνει πάρα πολλά προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω πραγματικά να σημειώσουμε τώρα πλέον πραγματική πρόοδο. Ελπίζω να το κάνουμε και στο πλαίσιο της πρότασης που έχουμε ενώπιόν μας. Πολύ επίσης αναφέρατε το θέμα της χρηματοδότησης, ε, το οποίο είναι βέβαια ένα ε, κεντρικό ζήτημα και όπως γνωρίζετε το ευρύτερο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα, θα είναι και πάλι αντικείμενο διαπραγματεύσεων ε, και πέρα από τις δικέ μου αρμοδιότητες και πέρα από τις δικέ σας αρμοδιότητες. Αυτό όμω που μπορούμε να κάνουμε είναι αν ε, η συζήτηση αυτή γίνεται να συνδεθεί με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, πού θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα επενδύσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αηφόρος ανάπτυξη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να μην βλέπουμε σιγά σιγά άλλες ε, περιφέρειες του κόσμου να μας ξεπερνούν. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα όσον αφορά τα, τη γενική χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Επίσης, αυτό μας φέρνει και στη συζήτηση της προσπάθειας ε, μεγαλύτερη σύνδεση ε, με τη συνοχή, με τα διαρθρωτικά και περιφερειακά ταμεία, με την ε, κοινή γεωργική πολιτική και με ε, πολιτικές που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γενικότερα. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένους στόχους και έχουμε καλέσει και τον Επίτροπο Χάν να είναι μαζί μας ε, στην ανεπίσημη συνάντηση που θα έχουμε στην Κοπενχάγη για να έχουμε μια πρώτη συζήτηση ήδη για το πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα, να ε, γίνει αυτή η σύνδεση που πρέπει να γίνει και να διαρθρώσουμε το διάλογό μας ε, ώστε να μπορέσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τις συμπεριλάβουμε στην προσπάθεια αυτή. Πολλοί εξημών συμφωνούν ε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διασύνδεση όλων αυτών των πολιτικών και ε, συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη αυτή. Θα προσπαθήσω να το επιτύχω. Πολλοί ε, εξημών μιλήσατε και για τη συζήτηση που γίνεται για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι γνωρίζουμε τη συζήτηση αυτή και τα ε, σημεία που θέσατε, γιατί έχουν τεθεί όχι μόνο από εσά, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις που είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη προγραμματική περίοδο ε, θα το συζητήσουμε και στην Κοπενχάγη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στο γεγονός ότι αν έχουμε αυτή την προσέγγιση που ε, επικεντρώνεται στις προκλήσεις και τις κοινωνικές προκλήσεις ιδιαίτερα, ε, πρέπει, αυτό μας βοηθά να έχουμε μια πολυτομεακή προσέγγιση και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε καλύτερη επαφή και με την αγορά με την εμπορευματοποίηση γιατί είναι πολύ σημαντικό οι αγορές και τα προϊόντα αντικατοπτρίζουν και την ανθρώπινη συμπεριφορά και γι' αυτό ακριβώς οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες έχουν πολλά να μας προσφέρουν από αυτού. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που κάποιοι από τους ε, ε, ε, ε από τους υπεύθυνους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης επιζητούν ακριβώς αυτό, ε, μια πολυτομεακή προσέγγιση και γι' αυτό ακριβώς είναι κάτι που πρέπει να το συμπεριλάβουμε στην όλη διαδικασία. Όμως δεν σημαίνει ότι μόνο ε, θα επικεντρωθούμε ε, στις κοινωνικές προκλήσεις ή μόνο σε μια πολετομιακή προσέγγιση. Μπορούμε να κάνουμε και τα δύο εκ παραλίλου. Νομίζω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Γιωχάνσεν και άλλοι συνάδελφοί σας να μην επικεντρωθούμε μόνο ε, στη χρηματοδότηση, δηλαδή υπό τους όρους ε, του πόσο προπολογισμό μπορούμε να έχουμε, αλλά και τι ε, αποτέλεσμα θα έχει ο προπολογισμός αυτός. Έχουμε πολλά μέσα ε, πώς μπορούμε να πετύχουμε το συντονισμό σε, μεταξύ εθνικού και κοινού ευρωπαϊκού επίπεδου και να υπάρχει και καλύτερη, ε, καλύτερος συντονισμός μεταξύ του τι συμβαίνει στα ερευνητικά Ινστιτούτα και στους διάφορους κλάδους. Νομίζω ότι πρέπει να καταφέρουμε να γεφυρώσουμε αυτά τα χάσματα γιατί ε, βρισκόμαστε μέσω, μέσω κρίσης και γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτήν την κοινή ευθύνη να ε, εξασφαλίζουμε ότι ό,τι χρήματα δαπανώνται, δαπανώνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Όσον αφορά τώρα τη συζήτηση για τις προκλήσεις, ε, πόσο ευρέως είναι ορισμένες οι προκλήσεις αυτές, ε, ετέθη αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι έχει να κάνει και με αυτό που ο κύριος Ρόλης στο τέλος. Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στις προκλήσεις αυτές Ω ευρύτερε προκλήσει ε, και χρειάζεται και πάλι μια πολυτομεακή προσέγγιση. Είναι επίση πολύ σημαντικό να μην καταλήξουμε σε, μια τόσο, σε ένα τόσο ευρύ ορισμό και σε ένα τόσο ευρύ κατάλογο που τελικά δεν επιτρέπει καμία ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Πρέπει να βρούμε αυτήν την λεπτή ισορροπία πρέπει να δώσουμε ενδεχομένω κάποιε προτεραιότητε σε κάποιε από τι κοινωνικέ προκλήσει. Το προτείνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνώ ότι ε, πρέπει ο ορισμός να μην είναι πάρα πολύ στενός αλλά ούτε και πάρα πολύ ευρύς και να μην αφήσουμε απ' έξω ε, ε, τομείς γνώσεων ή επιχειρήσεις που θα θέλαμε να συμμετέχουν. Συμφωνώ ε, με όσα είπατε για, την επιλογή, για τις επιλογές που πρέπει να κάνουμε. όσον αφορά την κινητικότητα και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Εγώ είμαι υπέρ ε, ότι, του ότι η γνώση πρέπει να είναι η πέμπτη ελευθερία που πρέπει να εξασφαλίσουμε η γνώση και οι ερευνητές πρέπει να μπορούν να ε, μετακινούνται και να εργάζονται ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ενισχύσουμε τα προγράμματα κινητικότητας ε, και περιμένω εναγωνίως τη συμμετοχή μου τη Δευτέρα στη διαβούλευση που έχει δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη συζήτηση αυτή. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος και στον συγκεκριμένο τομέα. Ο κύριος Ρόλ επίσης αναφέρθηκε στις παραδοσιακές ε, βιομηχανίες ε, σε σχέση με την πράσινη τεχνολογία. Σε αντιπαραβολή μάλλον με την πράσινη τεχνολογία. Πράγματι, είναι μια πρόκληση να έχουμε όσο το δυνατόν πιο αηφόρο ενέργεια, λιγότερα ορυκτά καύσιμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γυρνάμε την πλάτη σε παραδοσιακή βιομηχανία. Η παραδοσιακή βιομηχανία συχνά βρίσκει τρόπο να ανανεωθεί συμμετέχοντας στη συζήτηση αυτή. Αυτή είναι μια πρόκληση που θα εξακολουθεί να υφίσταται είτε εμείς την αντιμετωπίσουμε είτε όχι ε, και πολλές από τις καινοτομίες οι οποίες πρέπει να, να, να προβούμε ε, θα γίνουν πράγματι στο πλαίσιο της παραδοσιακής βιομηχανίας. Να σας πω ένα παράδειγμα, θα γίνει μια συζήτηση ε, για την ε, ε, τεχνολογία των βιολογικών προϊόντων το, την Άνοιξη. Και είναι ένας τομέας για τον οποίο υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες στο πλαίσιο του πράσινου τομέα και στο πλαίσιο της συζήτησης για την πράσινη ενέργεια. Δεν θέλω λοιπόν να δημιουργηθεί μία ε, αντιπαραβολή χωρίς να υπάρχει λόγος ε, μεταξύ πράσινης τεχνολογίας και παραδοσιακής βιομηχανίας. Ενδεχομένως να μην, είχα, να μην κάλυψα όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ε, ούτως ή άλλως θα επανέλθω στην επιτροπή σας τουλάχιστον τον νωρίτερο την Άνοιξη, όταν θα κάνουμε τη συζήτηση για το σεμινάριο, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συζήτηση και θα ήθελα να συμφωνήσω με όλους όσους είπαν ότι είναι μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή. Πρέπει να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας, είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε στο μέλλον και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση σε σχέση με την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ε, αφήνοντας πίσω την απώλεια θέσεων απασχόλησης. Οι αποφάσεις λοιπόν που θα λάβουμε στο πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας πρέπει να είναι ε, καρποφόρες, πρέπει να καρποφορήσουν ε, τουλάχιστον μακρο, μακροπρόθεσμα. Ελπίζουμε λοιπόν να μας βοηθήσετε να εξέλθουμε της κρίσεως και να περάσουμε σε μια, πιο, ε, σε μια περίοδο μεγαλύτερης ευημερίας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον Υπουργό για την παρουσία του, για τη σαφήνεια ε, και τη διάθεσή του να μας ε, ακούσει και για να ολοκληρώσουμε εδώ τη συνεδρία να σας πω ότι θα συνεχίσουμε στις 3 με τη μικρή ακρόαση για την ενεργειακή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ και ε, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Υπουργό. Είστε επανειδή.